Σύμφωνα με την μέσα διάταξη, ακολουθούν ψηφοφορίες. Επτά προτάσεις ψηφίσματος με θέμα την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη πρόταση ψηφίσματος είναι κοινή από τρεις πολιτικές ομάδες. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ε, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές και ε, η ΕΦΤΕ, Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία και αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα ψηφίσματα ε, των ομάδων αυτών. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα χωρίς τροπολογίες η πρόταση. Se han votado todos, se cierra. Ψηφίσατε όλοι. Vean, señorías, que... Bien. Se... Λοιπόν, πέρασε, είπαμε ψήφισαν 644, 297 υπέρ, 322 κατά, 25 εποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όπου δεν υπάρχει καμία τροπολογία. Sí. Θα ήθελα βάσει του άρθρου 157 του ιστορικού μας κανονισμού να μιλήσω για την τροπολογία υπαριθμού 2 του ΕΛΚ για το κοινό ψήφισμα για την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τροπολογία μου προκαλεί αποτροπιασμό. Δεν πρέπει να τη συζητήσουμε ούτε και να την ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Είναι ένα πυροτέχνημα αυτή η τροπολογία. Και γνωρίζουμε ε, εξάλλου τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Ε, Ο συντάκτης της τροπολογίας ε, καταδεικνύει την έλλειψη ανοχής ε, που έχει ε, και καταδεικνύει ότι επιθυμεί να κάνει μία ιερά εξέδαση και καταφέρεται κατά τον Νόμπελ που αποποιήθηκε την πορτογαλική υπηκότητα. Ευχαριστώ. Εντάξει, περνάμε στη σοφοφορία έχει ζητήσει το έλκονομαστική ονομαστική ψηφοφορία, απέσυρε το αίτημα και θα ψηφίσουμε διανατάσεως χειρός. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία θα ελέξουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Σε cierra votación. Ε, πέρας. 678 ψήφισαν, 258 υπέρ, 347 κατά. 73 αποχές. Απορρίφτεται Ακολουθεί η πρόταση ψηφίσματος ε, της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Χωρίς τροπολογίες έχει αποσυρθεί το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε δυνατά στους χειρός. Ψήφι υπέρ κατά αποχές Θέλετε επαλήθευση. Πολύ ωραία. Ας ελέγξουμε. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε cierra votación. Πέρασε. ψήφισαν 678, 301 υπέρ, 359, 51 ε, συγγνώμη, κατά, 26 αποχές, απορρίφτεται. Καλώς. Περνούμε τώρα. Ο κύριος Σασόλη. Πρόεδρε, ε, βάσει του άρθρου 147, σας υπενθυμίζω ότι στη συζήτηση που έγινε το 2007 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο αποφασίστηκε κατά να ε, μην ε, ισχύει αυτό για ε, ανθρώπους με υψηλά εξιώματα και αυτό το λέω για τις τροπολογίες του ΕΛΚ Μιλάμε για τον Τζόρτζο Ναπολιτάνο, τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σασόλη. Κύριε Σασόλη, μας λέτε ότι δεν είναι παραδεκτή αυτή η πρόταση βάσει του άρθρου 157 λέτε του κανονισμού μας. Συνεπώς η Προεδρία, ο Πρόεδρος Μπούζεκ εξέτασε το θέμα αυτό σε κάθε λεπτομέρεια, όπως μπορείτε να φανταστείτε και να κατανοήσετε. Και η ανάλυση του βασίστηκε στα εξής σημεία. Οι τροπολογίες 7, 8 και 9, στις οποίες εσείς ε, αναφέρεστε ή υπενήσεστε, έχουν άμεση σχέση με το κείμενο που τροποποιούν. Στη συνέχεια, δεν ζητούν απάλληψη ούτε αντικατάσταση ε, του συνόλου του κειμένου, ούτε τροποποιούν πολλές παραγράφους του κειμένου, ούτε αφορούν όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Συνεπώς, βάσει ε, της αυστηρής εφαρμογής των όσων ορίζει το άρθρο 157, ο πρόεδρος θεωρεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις έτσι ώστε οι τροπολογίες αυτές να μην μπορούν να θεωρούνται μη παραδεκτές. Άρα ο πρόεδρος αποφασίζει ότι ε, γίνονται δεκτές και τίθεται ε, σε ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά την αναφορά στον πρόεδρο ε, ε, Ναπολιτάνο, πρώην συνάδελφο και πολύ αγαπητό μας, τα προηγούμενα που υπάρχουν μας επιτρέπουν να συμπεριλαμβάνουμε ονόματα προσώπων πολιτικών στα κείμενά μας. Χωρίς καμία αμφιβολία, για να δώσουμε συνέχεια στο έτοιμά σας κύριε Σασόλη, ε, υπάρχουν και άλλοι ε, τρόποι και άλλοι διεύλοι ε, εκτός από το κανονισμό. Για παράδειγμα η προφορική τροπολογία ή καταψήφιση των τροπολογιών αυτών ακόμα. Καλώς. Sí. Señor Mauro, tiene usted... Κύριε Μάουρο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτω με την ερμηνεία τη Προεδρία για τι τροπολογίε. Όμω, έχω μια πρόταση προφορική τροπολογία. Α διατηρήσουμε όλε τι τροπολογίε και απλώ α απαλείψουμε το όνομα και το επίθετο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η πρότασή μου είναι λοιπόν σεβόμενη τη συνήθεια τακτική να μην έχουμε μνήες σε ονόματα και πρόσωπα, να αφαιρέσουμε την ανωνυμία του Τζόρτζο Ναπολιτάνο, αφήνοντα τη δυνατότητα να ψηφιστούν οι ίδιε τροπολογίε και τα κείμενά του. Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει το σεβασμό που έχουμε για την προσωπικότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που αντικειμενικά έκανε κάποιες δηλώσεις, παρέστη στη συζήτηση όλων των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο. Το λόγο ζήτησε ο κύριο Ρινάλντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω το κατά πόσο είναι αποδεκτέ τροπολογίε κατά την άποψη του Προεδρείου. Θα ζητήσω απλώ από του συντάκτε των τροπολογιών να σκεφτούν την πολιτική σκοπιμότητα του να τι ε, αποσύρουν. Δεν νομίζω ότι το να μην αναφερθεί το όνομα και το επίθετο του Πρόεδρου τη Δημοκρατία θα αλλάξει πολλά. Δεδομένου ότι ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία αναφέρεται σαφώ στις τροπολογίε αυτές. Νομίζω ότι είναι σχεδόν ε, τετουργία της δικής μας ε, νομοθετικής δουλειάς. Δεν φαντάζομαι στις τροπολογίες τους να αναφέρονται η βασίλισσα της Αγγλίας ή ο πρόεδρος της της Γερμανίας σε ανάλογες τροπολογίες άλλων νομοθετικών σωμάτων. Θα έλεγα λοιπόν να αποσυρθούν οι τροπολογίες 7, 8 και 9 από το ψήφισμα. Πολύ ωραία. Ε, Κύριε Σασόλη δεδομένου ότι εσείς θέσατε αυτό το ζήτημα και ακούσαμε μία πρόταση του κυρίου Μάουρο απαντώντας τη δικιά σας θέλετε να λάβετε το λόγο για να απαντήσετε Είμαστε υπέρ της απάλληψης του ονόματος και επιθέτου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μας για τις τροπολογίες αυτές βεβαίως δεν θα ψηφίσουμε υπέρ Συνεπώς, αφαιρείται η ονομαστική αναφορά το όνομα τεπώνυμο του αρχηγού του Ιταλικού κράτους, του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Έχουμε πρόταση ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων, σοσιαλιστές και δημοκράτες, φιλελεύθεροι, πράσινοι και ενωτικοί αριστερά, που αντικαθιστά όλες τις ε, προηγούμενες προτάσεις ψηφισμάτων των ομάδων αυτών. Η τροπολογία παριθμών 5. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 10 με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Περάσα. 687 ψήφισαν, 306 υπέρ, 343 κατά 38 εποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 8 με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εψήφισαν 676, 318 υπέρ, 343 κατά, 15 εποχές απορρίπτεται. Καλώς, τώρα λοιπόν έχουμε μια προφορική τροπολογία του κυρίου Μέλλο. Έχετε το λόγο. E Πρόεδρε, προφορική τροπολογία είναι εξή. Λυπούμαστε και εκφράζουμε τη θλίψη μας για τις επιπτώσεις από την σοσιαλιστική κυβέρνηση της Πορτογαλίας που οδήγησαν στην απόφαση να κλείσει η εφημερίδα και το τουριστικό κανάλι TV και καταγράφει ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να γίνει αντικείμενο έρευνας από την ε, ε, Πορτογαλική Ρυθμιστική Αρχή. Σας ευχαριστώ κύριε Μελό. Διαφωνεί κανένας βουλευτής με την έγκριση αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται παραδεκτή η προφορική τροπολογία. Ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την παράγραφο υπαριθμών 3, παρακαλώ. Σε Εψήφισαν 677, 338 υπέρ, 320 κατά, 19 αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε την παράγραφο 4 με ονομαστική πάλι ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. Ε, ψήφισαν 686. 331 υπέρ, 326 κατά, 21 αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 6 με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. 687 ψήφισαν, 301 είπε, 368 κατά, 18 αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα ονομαστικά την παράγραφο 5, αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 686 ψήφισαν, 345 υπέρ, 324 κατά, 17 αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 6, αρχίζει η νομιστική ψηφοφορία. 684 ψήφισαν, 342 υπέρ, 327 κατά, 15 αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 7 με ονομαστική και πάλι ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. Εψήφισαν 687, 346 υπέρ, 318 κατά, 23 αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την Παύλα υπαριθμών 7 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εψήφισαν 687, 345 υπέρ, 323 κατά, 19 αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 7. Ονομαστικά αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε cierra 688, 302 υπέρ, 346 κατά, 40 αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 9. Ονομαστική ψηφοφορία. Se cierra la votación. Πέρας. 683 ψήφισαν, 326 υπέρ, 335 κατά. 22 εποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την αιτιολογική σκέψη Β. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά χρειάζεται επαλήθευση. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Ψήφισαν 688, 343 υπέρ, 326 κατά, 19 αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 2 με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε στι 690. 269 υπέρ, 338 κατά, 83 αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε τροπολογία υπέρ 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται υπερθυμό 3. Τώρα, σε δύο τμήματα έχουμε την αιτιολογική σκέψη γάμα, ε, λατινικό. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα πρώτα, ε, Κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, ονομαστικά παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας ψήφισαν 689, 331, 39 συγγνώμη, υπέρ, 331 κατά 19 αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα τροπολογία υπαριθμών 1 με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Σε θεία Πέρας. Εψήφισαν 691, 271 υπέρ, 339 κατά, 81 αποχές. Απορρίφτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την αιτιολογική σκέψη D. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Αποχή εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. Ψήφισαν 688, 261 είπε 338 κατά, 89 αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε μια προφορική τροπολογία του κυρίου Σάχερ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα το ότι δεν θα έπρεπε να δεχτεί το Κοινοβούλιο ψηφίσματα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παραθέτω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, την Ουγγαρία. Ο Υπουργός Οικονομικών κίνησε δίωξη κατά ενός δημοσιογράφου γιατί δεν του άρεσαν τα άρθρα του, τα οποία ήταν κατά αυτού. Οπότε μιλάμε εδώ για έναν πρωθυπουργό που κινεί ποινική δίωξη κατά των δημοσιογράφων. Νομίζω το πρόβλημα όπως και στην Ουγγαρία είναι ότι εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, καλό τους συναδέλφους να μην υπερψηφίσουν αυτή την τροπολογία γιατί ε, έτσι ξεκάθαρα θα φανεί ότι πρόκειται για ένα υπερθέαμα εδώ για να τρομάξουμε τον Πρωθυπουργό μιας χώρας επειδή και μόνο η κυβέρνηση δεν είναι από τη δική σας πολιτική οικογένεια. Αλλά όταν μιλάμε για σοσιαλιστική κυβέρνηση ακολουθούνται άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχθεί αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά για να ασκηθούν πιέσει ε, σε δημοσιογράφου που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθορά ε, όπου ε, καταφέρονται κατά των πρωθυπουργών και άλλων υψηλών αξιωματούχων. Μιλώ για τον κύριο Τόμας Μπίντροχ, κυρίως για τον δημοσιογράφο Μπόντρα Χίλοπ η ποινική δίωξη κινήθηκε κατά του δημοσιογράφου που διερευνούσε ένα σκάνδαλο που εμπλεκόταν ένας ψηλός αξιωματούχος της κυβέρνησης ε, και ένα από τα μέλη του επιτελείου ενός Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Ασκείται μεγάλη πολιτική πίεση στο δημοσιογράφο αυτό στην ε, Ουγγαρία. Ε, καταψηφίστε αυτή την τροπολογία για να παραμείνει αξιόπιστο το κοινοβούλιο για να δείξετε ότι δεν εκφοβίζετε κάποιον που απλώς δεν σας αρέσει και ότι πραγματικά είστε υπέρ ε, της ε, ελευθερίας του τύπου στην ε, Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σάγερ για την προφορική σας τροπολογία αναγνώστηκε. Κάποιος βουλευτής διαφωνεί με την προφορική τροπολογία του κύριου Σάγερ. Σας παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία, κυρίες και κύριοι. Silencio. Ησυχία, παρακαλώ. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε. Ακούσαμε την τροπολογία του κύριου Σάγερ, η οποία απεριφθεί. Ψηφίσουμε τώρα την αιτιολογική σκέψη ε με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Ψήφισαν 684. 331 υπέρ. 327 κατά. 26 εποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 11. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Σε cierra Πέρας. Εψήφισαν 689, 319 υπέρ, 344 κατά, 26 αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνορο της πρότασης ψηφίσματος, της κοινή πρότασης, με ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει. Se cierra la votación. Πέρα. 686. 335 υπέρ. 338 κατά. 13 αποχές.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 Κύριε Μάουρο, καθίστε κάτω. Λοιπόν, περνούμε τώρα στην εξέταση της πρότασης ψηφίσματος της ομάδας των Πρασίνων και της ε, Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας χωρίς καμία τροπολογία. Συγγνώμη. Ε, ψήφι υπέρ. κατά Vamos a Έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Σε Πέρασε. 675 ψήφισαν. 321 είπε. 346 κατά 8 αποχές απορρίψετε. Και στη συνέχεια τώρα θα ψηφίσουμε την ε, πρόταση ψηφίσματος της Ευρώπης για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία χωρίς τροπολογίες ψηφιπέ. Κατά. Αποχές Αρχή ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Πέρας. 676 ψήφισαν, 257 υπέρ, 399 κατά, 20 εποχές απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Ανατικής Αριστεράς και Βόρειας Πράσινης Αριστεράς χωρίς τροπολογίες ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ψηφίζουμε την πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών, χωρίς τροπολογίες. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. αρχής τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 683 σε ψήφισαν. 333 υπέρ, 345 κατά και 5 εποχές. Απορρίπτεται. Και τελευταίο ψήφισμα, έχουμε και άλλο. Είναι η πρόταση ψηφίσματος των φιλελευθέρων. Χωρίς τροπολογίες και αυτή. Ε, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Σε Πέρας. Εψήφισαν 684. 338 υπέρ. 338 κατά.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 Πρόεδρε, για να σας ενημερώσω, ζητώ το λόγο, για κάτι πολύ σοβαρό που δεν έχει να κάνει με την ψηφοφορία μας. Ζητώ από την Προεδρία του Κοινοβουλίου άμεσα να αναλάβει δράση ενημερωτική. Να βεβαιωθούμε ότι οι δικές μας ασυλίες και τα προνόμια θα διασφαλιστούν, διότι σήμερα ένας βουλευτής από την αντιπροσωπεία μας, σήμερα το πρωί κιόλας, δέχτηκε την έφοδο στην ιδιωτική του κατοικία από αστυνόμους ε, της Ιταλικής αστυνομίας στο Στρασβούργο και άμεσα απομακρύνθηκε από το Στρασβούργο με την πρωτοβουλία της ε, δικαστικής εξουσίας της Ιταλίας η οποία διέθετε το ένταλμα για ε, Ιταλό βουλευτή. Μπήκε στην ιδιωτική του κατοικία λοιπόν και αυτό έχει άμεση σχέση με τι δικέ μα ασυλίε και δικαιώματα. Ζητώ λοιπόν απλώ από το Κοινοβούλιο αυτό και από την Προεδρία να, λάβει δράση, να αναλάβει δράση, να βεβαιωθεί ότι η αστυνομία και η δικαστική εξουσία τη Ιταλία ε, κατά του κυρίου Μαστέλα ε, αν ήταν μέσα στα πλαίσια του σεβασμού του δικαίου και των ε, χαρακτηριστικών των χαρακτηριστικών των ασυλιών και προνομίων μας. Η Προεδρία θα δώσει συνέχεια στο θέμα αυτό και θα το διερευνήσει για να υπερασπιστεί χωρίς καμία αμφιβολία τα προνόμια και τις ασυλίες μας. Κύριε Λαντσμπέργκης. Κύριε Λαντσμπέργκης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω η προηγούμενη ατυχής ψηφοφορία για ένα λιθουανικό νόμο στην ανύπαρκτη ακόμα εκδοχή του αυτή η ατυχής λέω ψηφοφορία ελπίζω να βοήθησε πολλούς συναδέλφους να καταλάβουν ποιος είναι ο κίνδυνος και θα πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταντήσει η Σοβιετική Ένωση Ευχαριστούμε κύριε Λαντσμπέργης. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Και το λόγο έχει ο κύριος Ριμπελίνη. Κύριε Ριμπελίνη, έχετε το λόγο.